Και πηγαίνουμε τώρα στις παρεμβάσεις διαρκείας ενός λεπτού. Πρώτη, η κυρία Κλούνε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στις 25 Νοεμβρίου είναι η Διεθνής ημέρα για την πάταξη της βίας κατά των γυναικών που είναι τα πρώτα θύματα της οικιακής βίας, πολύ ασθενείς και ευάλωτες σε αυτή την κατάσταση. Να σας ενημερώσω λοιπόν ότι πρόσφατα το κράτος της Ιρλανδίας υπέγραψε τη σύμβαση της ε, Κωνσταντινούπολης ε, για την ε, επάταξη της βίας των γυναικών και της οικιακής βίας. Η οικιακή βία συχνά θεωρείται ότι πρέπει να μείνει πίσω από τις κλειστές πόρτες του σπιτιού όμως. Αυτό πρέπει να αλλάξει και πρέπει να δώσουμε έμφαση στην υποστήριξη στις γυναίκες και στη δημοσιοποίηση. Δεν έχουμε μόνο τη σωματική βία αλλά και την κακοποίηση ψυχολογικής φύσεων, φύσεως η οποία είναι ακόμα πιο δύσκολη. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των γυναικών στην Ευρώπη κάθε μέρα αντιμετωπίζουν βία. Το νομικό, πολιτικό και αστυνομικό σύστημα πρέπει να εκπαιδευτούν ώστε να αναγνωρίζουν τη βία αυτή και να μην τη θεωρούν κάτι που πρέπει να παραμείνει στο σπίτι. Πρέπει να υποστηριχτούν τα θύματα και οι θύτες να γνωρίζουν τις επιπτώσεις της κατάστασης αυτής. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω την ανησυχία της χώρας μου και των συμπολιτών μου εξαιτίας της ε, κλιμάκωσης της ε, βίας ε, και του φόβου των παιδιών που ζουν στις άλλες χώρες. Θεωρώ ότι η ασφάλεια των πολιτών στην Ευρώπη είναι κέριο ζήτημα. Νομίζω ότι ως πρόεδρος, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου πρέπει να έρθουν εδώ στο Κοινοβούλιο και να παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους για τη μετανάστευση τους πρόσφυγες, την ασφάλεια των συνόρων και των πολιτών της Ευρώπης γιατί ε, με τις ε, ποσοστώσεις δεν λύνουμε το θέμα. Μπορεί να έχουμε υψηλό βαθμό ε, συναγερμού για πολύ καιρό, να έχουμε απώλειες ζωής, αλλά το πρόβλημα δεν λύνεται. Δεν βγαίνουμε από την κρίση. Θέλουμε μια ασφαλή Ευρωπαϊκή Ένωση με ίση μεταχείριση. Δεν θέλουμε μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων και έλλειψη ασφάλειας. Όλοι έχουμε υπογράψει τις ίδιες συνθήκες και πρέπει όλοι να αντιμετωπιζόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Πατήξ Φορστρόχ, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, με τα ανοιχτά σύνορα, την τρομοκρατία και την νομοθεσία σχετικά με το θέμα αυτό ε, πρέπει να συζητήσουμε και να συνδέσουμε τα θέματα. Οι ε, πράσινοι και αριστεροί θεωρούν ότι τώρα έχουμε μεγαλύτερη ευθύνη για, λόγω της παρακολούθησης των πολιτών. Όμως βλέπετε ότι έχουν επανέλθει οι συνοριακοί Έλεγχη. Φαίνεται ότι ο τρόμος ε, είναι εκεί και όλους ε, μας ε, τρομάζει. Οι τρομοκράτες έχουν αυτή τη στιγμή φέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των νόμιμων όπλων της οπλοφορίας. Είναι ζητήματα τα οποία έχουν αρχίσει να συζητούνται. Επίση πρέπει να ελέγχουμε τα σύνορα. Το Τσέσου και η κυρία Ρολ Ρολμάγερ δεν το θέλουν. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα. Για να τόμ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι με πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση ο πόλεμος για τη Συρία και είναι επικείμενη απειλή. Ε, είδαμε τις τρομοκρατικές επιθέσεις ε, στο Παρίσι και αυτό είναι απόδειξη ότι έφτασε ο πόλεμος ε, στην Ευρώπη. Μετά τις ενέργειες επιθέσεις της Ρωσία στη Συρία άλλαξε η κατάσταση και θα πρέπει να δούμε τελικά ε, κερδίζει έδαφος ε, το Ισλαμικό κράτος ε, έχει γίνει μια, κατά κάποιο τρόπο μια εναλλακτική λύση για την, σε σχέση με την Δυτική Συμμαχία και αμφισβητείται ο ρόλος της Ρωσίας σε αυτό το συνασπισμό. Ε, είναι λαθασμένη η προσέγγιση που φέρνει την, το διχασμό στα πλαίσια της... Ε, Ο πόλεμος κατά του Ισλαμικού κράτους είναι πάρα πολύ σημαντικός και θα πρέπει για να εξυπηρετήσουμε γεωπολιτικά συμφέροντα να επιτρέψουμε να υπάρξει ε, διχογνωμία σε σχέση με τον, το δυτικό συνασπισμό κατά του Ισλαμικού κράτους. Ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κατάσταση των ε, μεταναστών και προσφύγων στα Δυτικά Βαλκάνια, σε αυτή τη μαζική ροή προσφύγων και μεταναστών, μας οδηγεί σε μια παράδεκτη κατάσταση από ανθρωπιστικής πλευράς. Επιδεινώνεται η κατάσταση τις τελευταίες ημέρες με την ανύψωση παράνομων τυχών και ε, κλείσιμο συνόρων από πλευρά ε, κρατών μελών που δικαιολογούνται που δεν δικαιολογούνται σε καμία περίπτωση διότι πρόκειται για ευπαθή άτομα σε απόγνωση ε, και δεν μπορούμε να τους γυρίσουμε την πλάτη. Χρειαζόμαστε μια κοινή απάντηση, μια κοινή απόκριση που θα βασίζεται στις κοινέ αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, τις αξίες που προκυρήσει αλλά δεν εφαρμόσει ε, για να προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους από το χάος και από τον πόλεμο που τροφοδότησε ή και προκάλεσε η Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, χρειαζόμαστε νόμιμες οδούς μετανάστευσης ε, και ε, θα πρέπει να σταματήσουμε αυτή την κατασταλτική διακριτική μεταχείριση κατά των προσφύγων και την βία που διαπιστώνουμε στα σύνορα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι φιλικά κέντρα υποδοχής για τους μετανάστες και πρόσφυγες. Ευχαριστούμε, Χόρδη Σεβάστιν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εμβληματική η μέρα του Νοεμβρίου για αυτούς που διεκδικούν την φασιστική δικτατορία του Φράνκο. Σε πολλές πόλεις έγιναν εκδηλώσεις υπέρ του καθεστώτος Φράνκο και στο Αλικάντε όπου το 77 σκοτώθηκε ο Μιγγέλ Γράου από έναν υποστηρικτή του φασισμού που μετά έλαβε αμνηστία. Πρόκειται για μια συνέχιση της ατιμωρησίας και προσβολή της ιστορικής μνήμης. Η τα θύματα της δικτατορίας αυτής ε, που δολοφονήθηκαν δεν την χάνουν της απαραίτητης ε, προστασίας. Η κυρία Ρέντινγκ λέει ότι και σωστά ότι δεν μπορεί να μείνει σιωπηλή ενώπιον της τάσης ενός ε, κράτους μέλους προς τον, ε, προς ολοκληρωτισμό. Πρέπει να δώσουμε απαντήσεις και να ζητήσουμε από το Ισπανικό κράτος να υποστηρίξει τα δεοντολογικά και τις νόμιμες υποχρεώσεις. Ευχαριστώ. κυρία δεν έχει το λόγο. Τώρα, ευχαριστώ. Οι χριστιανοί είναι αυτοί που κυνηγούνται περισσότερο από παντού στον κόσμο. Πολλοί από αυτούς στη Μέση Ανατολή. Για αιώνε στη Μέση Ανατολή ζήσαν, προσευχή, ζούσαν, προσεύχονταν και δούλευαν χριστιανοί. Από την κατάρριψη ωστόσο των κοσμικών ηγετών στην περιοχή, η ISIS ξεκίνησε μία καμπάνια κατά του χριστιανισμού λαιλατούνται και καταστρέφονται αρχαίες εκκλησίες. Ε, χριστιανές κοπέλες πολλούνται σε σκλαβοπάζαρα ε, σεξ, ενώ οι χριστιανοί όπου επιβιώνουν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Βλέπουμε να πετάνε από τις στέγες ομοφιλόφιλους και η ε, σιωπή τόσων ομάδων, ε, τόσων πολλών ομάδων ε, υποστηρικτών της ομοφιλοφιλίας είναι εκοφαντική. Ο εξτρεμισμός φτάνει και στη χώρα μου αυτή τη στιγμή. Οι ομοφιλόφιλοι άντρες και γυναίκες ε, αντιμετωπίζονται διακριτικά από ριζοσπαστικές ομάδες. Αυτό είναι απαράδεκτο. Η περιοχή του Ανατολικού Λονδίνου είναι μια επικίνδυνη περιοχή για τους γκέι άνδρες. Ελπίζω αυτός που θα κερδίσει το Λονδίνο, τις εκλογές του Δήμου του Λονδίνου να αντιμετωπίσει σαν προτεραιότητα αυτό. Η κυρία, ο κύριος Κοράου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το PSR 2009-10 οδήγησε σε εκατοντάδες ε, οδήγησε εκατοντάδες ε, εργαζόμενους να εγκαταληφθούν αφού απογοητεύθηκαν. Αυτό που περιγράφω είναι ένα αποκαλυπτικό σενάριο που συμβαίνει στην περιοχή μου, στη Σικελία, όπου γύρω στις 400 αγροτικές εκμεταλλεύσεις κινδυνεύουν να κλείσουν αν τα, οι, οι πόροι του PSR για το 2011-2013 ε, δεν προχωρήσουν. Πολλοί μου ζήτησαν να υπάρξει παράταση των πόρων αυτών. Μαζί με άλλους συναδέλφους από το κίνημα πέντε αστέρων ζητήσαμε να ασκήσουμε πίεση στις εθνικές και περιφερειακές αρχές. Ωστόσο τον τελικό λόγο τον έχει Επιτροπή. Ζητώ σήμερα από την Επιτροπή με ταπεινότητα να παρατείνει, να δώσει αυτή την παράταση που είναι ζωτική για τον κλάδο της γεωργίας ε, που είναι τόσο σημαντικός για την περιοχή μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κοράου. Η κυρία Ντομινίκ Μπίλντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ασθένεια του Αλσχαϊμέρ και συναφής ε, εκφυλιστικής ασθένειας πλήττουν 60 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη περίπου και ε, είναι αυξανόμενος ο αριθμός των περιπτώσεων. Στη Γαλλία 200.000 νέα κρούσματα ε, στην, υπάρχουν στη Γαλλία κάθε χρόνο και ένας στους τέσσερις έχει κάποιον στο οικογενειακό του περιβάλλον και τόσο ασθενής όσο και η οικογένεια και οι φίλοι του πλήττουν από αυτή την ασθένεια διότι ανακόπτονται βασικές πνευματικέ λειτουργίες, η μνήμη συγκεκριμένα και δεν υπάρχει προ το παρόν καμία θεραπεία για τη θεραπεία του Αλσχάμερ παρότι κάποιε θεραπευτικές αγωγές μπορούν να επιβραδύνουν τη διαδικασία. Είναι η πρώτη αιτία εξάρτησης ε, του ανθρώπου που χρειάζεται περίθαλψη και γι' αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα στην Ευρώπη 24 βουλευτές και υποφαινόμενοι διακομματικά υπογράψαμε ένα κοινό ψήφισμα για να ζητήσουμε αύξηση των κονδυλίων για την έρευνα. Είναι προτεραιότητα για μας. Θα καλούσα και όλους τους συναδέλφους να, να πάνε να ε, υπογράψουν αυτήν την δήλωσή μας. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε ήδη ακούσει πάρα πολλές ε, ομιλίες ε, για τα ε, τζαμπιά και για τον Ισλαμισμό εδώ. Να πω λοιπόν ότι υπάρχει ένα ερώτημα που τίθεται. Δεν θεωρούμε ότι κάπου τα πράγματα έχουν πάρει το λάθος δρόμο. Δεν θεωρούμε ότι Όταν έχουμε ε, ανθρώπους που μιλάνε για τα τζαμιά, δεν είναι αυτό μίσους, αλλά ε, ε, όταν κανείς πηγαίνει να επισκεφτεί τέτοιους χώρους, ε, στην ουσία τα βλέπει ως χώρους αξιοθέατα. Στο Παρίσι Κυρία Πάουνοβα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι άθλιες επιθέσεις στο Παρίσι αλλά σχεδόν και και τα θύματα του Σαρλί Εμπντό και οι 48 περασμένες ώρες στις Βρυξέλλες στην ουσία ένα πράγμα πρέπει να μας μάθουν ότι δεν μπορούμε πλέον να ζήσουμε στο φόβο και την ανασφάλεια Γι' αυτό μετά από δέκα μέρες από την ε, ε, τρομοκρατία στο Παρίσι σας λέω ότι δεν πρέπει να περιμένουμε τόσες μέρες όσες περιμέναμε μετά το Σαρλί Επτό, 300 μέρες και για να αντιδράσουμε. Πρέπει να ενισχύσουμε βασικά στοιχεία όπως τη Frontex, να την κάνουμε ένα πραγματικό φύλακα των εξωτερικών συνόρων και πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τους ριζοσπαστικούς ε, μαχητές μέσα στο έδαφος μας. Πρέπει να ε, βγάζουμε πληροφορίες και να τις μοιραζόμαστε, γιατί μια μέρα χωρίς αυτό ακόμα είναι μια μέρα χωρίς, με φόβο για τους πολίτες μας. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα... Η κυρία Βιωρίκα Ντάντσιλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με μεγάλη μου ανησυχία παρατηρώ ότι πρόσφατα Υπάρχει λόγος για την επαναφορά της Ευρώπης των δύο ταχυτήτων είναι ανησυχητικό γιατί ένας από τους ηγέτες της Ευρώπης, ο κύριος Γιούγκερ, ενθαρρύνει μια τέτοια ιδέα που είναι εναντίον των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βασίζονται στην συνοχή, στην απάλυση των διαφορών. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια και την ανεργία των νέων αν μειώσουμε την ένταξη, πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ε, υπερασπιστεί τον εαυτό της έναντι των εξωτερικών εχθρών αν οι ίδιοι οι ηγέτες της είναι διχασμένοι. Από το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν υπάρξει κλήσεις για να μειώσουμε τα δικαιώματα των μεταναστών. Όμως τώρα χρειαζόμαστε περισσότερη ανοχή και αλληλεγγύη και ενότητα. Ο πρόεδρος ε, της Κομισιόν πρέπει να έχει ως καθήκον να υποστηρίξει αυτά που λέει, γιατί εγώ δεν πιστεύω στην Ευρώπη των δύο ταχυτήτων και σε μια Ευρώπη που βασίζεται σε κάτι τέτοιο. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Νταντζίλα και τώρα Άγγελ Μπαμπάνσκι. Ευχαριστώ. Τα πρόσφατα τραγικά περιστατικά από τις επιθέσεις του Ισλαμικού κράτους ε, στην Ευρώπη είναι άλλο ένα ανα... αποδεκτικό στοιχείο για αυτά που ισχυριζόμαστε τα τελευταία χρόνια σε σχέση με την ε, ριζοσπαστικοποίηση στην Ευρώπη. Θα πρέπει να δράσει εσπεσμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση και να προστατεύσει τα σύνορά της. Τα σύνορα της Βουλγαρίας είναι τα μακρύτερα ε, εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήθελα να απευθυνθώ ε, στους συναδέλφους, ε, κυρίως από το ΕΛΚ, που θεωρούν εμάς υπεύθυνους ε, για την ανεύθυνη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει άμεσα να κλείσουν τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμπίπτουν με τα σύνορα της χώρας μου. Αμέσως αμελητή θα πρέπει να απελαθούν οι παρανόμως διαμένοντας άλλο δαπή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να εντοπιστούν οι τρομοκρατικοί οι πυρήνες ε, του Ισλαμικού κράτους ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να δράσουμε άμεσα. Δεν υπάρχει άλλος ε, τρόπος. Είναι μονόδρομος. Μόνο έτσι μπορούμε να σώσουμε τις χώρες μας. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπιλμπάου Μπαραντίκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα στην Ισπανία οι οικογένειες 100.000 περίπου ατόμων που έχουν εξαφανιστεί κατά τη διάρκεια της Φρανκικής ε, δικτατορία συνεχίζουν να ψάχνουν τους, ε, τους συγγενείς Αυτό δεν έχει υλοποιηθεί παρότι η υποστήριξη της, ε, του βασικού κόμματο τη αντιπολίτευση επιτρέπει να γίνει παραπομπή των ορισμένων ατόμων αυτών ατόμων από αυτά για τι τις αδικίες που είχαν γίνει στο παρελθόν. Αυτό δεν γίνεται ωστόσο λόγω της κυβέρνησης. Πρέπει τα θύματα να έχουν την ίδια αντιμετώπιση με άλλα θύματα ολοκληρωτικών καθεστώτων στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γουαρίστια Μπάουντς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο Δικαιωμάτων Ανθρωπτορία πολλές φορές μίλησαν κατά της άρνησης και της απλοποίησης των εγκλημάτων του φραγκισμού, ωστόσο καταγράφονται ακόμα και σήμερα στην Ευρώπη περιπτώσεις απαράδεκτες όπως ε, η συνεχιζόμενη πληρωμή από πλευράς Γερμανίας συντάξεων σε φραγκικούς εθελοντές της της μπλε ταξιαρχίας ή η προστασία από πλευράς της ισπανικής κυβέρνησης της ατιμορρησίας για τα εγκλήματα της δικτατορίας μέχρι και σήμερα. Είναι καιρός να αποκατασταθεί η αξιοπρέπεια, ο σεβασμός και η μνήμη για χιλιάδες οικογενειών που εδώ και δεκαετίες περιμένουν απαντήσεις και δικαιοσύνη. Τούτο απαιτεί συλλογικέ δεσμεύσεις και συμμετοχική διαδικασία, διότι η ιστορική μνήμη ανήκει σε όλους μας. Και το Κοινοβούλιο έχει και την ευθύνη να πει ξεκάθαρα ότι η ατιμορρησία δεν είναι δημοκρατία. Ενώπιον των εγκλημάτων του φρακισμού ζητούμε δικαιοσύνη και αποκατάσταση ευχαριστώ. Η κυρία Τιτσιάνα Μπεγκίν, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ και χρόνια η Κίνα, η Κίνα μας εισβάλλει με, ε, με φοβερά χαμηλής ποιότητας προϊόντα. Η συνένοχη αυτής της πολιτικής είναι εδώ. Από το Δεκέμβριο του 2016 η Κίνα θα χρησιμοποιηθεί ως οικονομία αγοράς και δεν μπορούμε να προστατεύουμε πλέον τα προϊόντα μας όπως τα κάνουμε τώρα. Ωστόσο η Κίνα δεν είναι οικονομία ανοιχτή αγοράς, δεν έχει καμία νομική παράμετρο τέτοια και δεν μπορεί να γίνεται η επιλογή αυτή από την Επιτροπή ένα όργανο που δεν εκλέγεται από κανέναν. Ξέρετε ότι πάνω από 3 εκατομμύρια θέσει εργασία στην Ευρώπη εξαρτώνται από τι επιλογέ αυτού του μη αιρετού οργανισμού. Η Ιταλική κυβέρνηση καταλαβαίνει ότι 700.000 θέσει εργασία στην Ιταλία και μόνο εξαρτώνται από την απόφαση αυτή. Βεβαίω και το γνωρίζει. Όλοι το ξέρουν. Όλοι σιωπούν ωστόσο. Ούτε καν ο Πρωθυπουργό μα. Στην Ιταλία κανεί δεν μιλάει για το θέμα αυτό πλην του, ε, του Υφυπουργού Καλέντο. Αλλά αυτό ε, δεν θα με εξέπληρε αν και αυτός ε, δεν σταμάτηγε να μιλήσει. Ίσως κανέναν ενδιαφέρον η θέση εργασίας. Ευχαριστώ. Συνάδελφε. Η κυρία Ρωμάνα Τόμσκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι μετανάστες έρχονται στην Ευρώπη και μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα πάνω από 250.000 μετανάστες ταξίδεψαν μέσω της Σλοβενίας που στην ουσία είναι πάνω από το 10% του συνολικού πληθυσμού και έγιναν αιτήσει ασύλου. Οι περισσότεροι από αυτούς τους μετανάστες όμως είναι οικονομικοί. Έρχονται οι περισσότεροι χωρίς έγγραφα. Είμαστε κομμάτι του Σέγγεν και εμείς πρέπει να προστατέψουμε τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αστυνομία της Σλοβενίας έχει ανοιχνεύσει πολλούς ε, μετανάστες που χρησιμοποιούν αυτές τις ροές δυστυχώς και πρέπει να αναρωτηθούμε κατά πόσο μπορούμε να εμπιστευτούμε τις υπηρεσίες ασφαλείας ε, και τις ικανότητες που έχουμε αν είναι ε, εκεί αυτές ε, οι υπηρεσίες και μετά από τις επιθέσεις στο Παρίσι πραγματικά με για την κοινή πολιτική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Jonás presidente. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα πρώτα μου λόγια σήμερα είναι για να εκφράσω φόρο τιμή στα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στην Ευρώπη, που δείχνουν την ανάγκη να έχουμε μια πολιτική άμυνας και ασφάλεια στην Ήπειρό μας. Θέλω να μιλήσω σήμερα για την συζήτηση για την δυνατότητα να δοθεί στην Κίνα όρο η συνθήκη της οικονομίας αγοράς κάτι που μπορεί να επηρεάσει ρητά και ξεκάθαρα τον, ε, τη βιομηχανία στην Ευρώπη, σημαντικού ε, τομεί ιδιαίτερα, τη χαλιβουργία για παράδειγμα, πολύ σημαντική για την Αστορία. Η κινέζικη οικονομία δεν είναι οικονομία αγορά. Ε, η πιστοτική πολιτική γίνεται από το κράτο η οποία που ζητά από τους εργαζόμενους να μετακινηθούν από τη μία περιοχή στην άλλη. Τι οικονομία αγορά είναι αυτή όταν υπάρχει έλεγχο τη πιστοτική πολιτική και των ανθρώπων. Αυτό δεν μπορεί να το ακολουθήσει η Ευρώπη γιατί έρχεται εις βάρος των βασικών αρχών της Ένωσης και επηρεάζει αρνητικά την περιοχή μου όπως την Αστουρία. Ο κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η μνημονιακή συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ψήφισε πριν μερικές μέρες ένα ακόμη επέσχυντο νόμο με προαπαιτούμενα που απαιτούσαν η τρόικα και οι δανειστέ. κύρια αιχμή του νόμου είναι τα κόκκινα δάνεια. οι αλλεπάλληλε ανακεφαλαιοποιήσεις που έγιναν θα έπρεπε ήδη να είχαν από καιρό διαγράψει πολλά κόκκινα δάνεια διότι έλαβαν για αυτό το σκοπό κεφάλαια. αντί γι' αυτό η εφαρμογή των ρυθμίσεων του συγκεκριμένου νόμου θα οδηγήσει σε δεκάδε χιλιάδε κατασχέσει και πληστηριασμό κατοικιών ελλήνων δανειοληπτών και τα διεθνή κερδοσκοπικά πιστωτικά ιδρύματα τα διάφορα φαντ και τα κοράκια θα βάλουν χέρι στα σπίτια των ελλήνων πολιτών. τέτοιο νόμο δεν είχαν καν τολμήσει να ψηφίσουν ούτε οι προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις. αυτό ακριβώς δυστυχώς ψήφισε η μνημονιακή συγκυβέρνηση σύριζα ανέλ. οι έλληνες πολίτες θα παλέψουμε ειρηνικά και δημοκρατικά και δεν θα επιτρέψουμε κανένα συμπατριώτης μας να χάσει το σπίτι του όπως συνέβη στην ισπανία. κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη κανένα σπίτι στα κοράκια. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σαδαβί, Σαμιένικ, Ιώρο Ράδος. Ευχαριστώ, πρόεδρε πολιτική ασφάλεια και η κοινή εξωτερική πολιτική υπάρχει εδώ και 20 χρόνια και η κοινή αμυντική πολιτική υπάρχει εδώ και 25 χρόνια και οι δύο πολιτικές ε, έχουν διαδοχικά διαφορετικά μέσα, διαφορετικούς τρόπους δράσης, διαφορετικά θεσμικά όργανα. Όμως για την ισχύ αυτών των πολιτικών δεν έχει σημειωθεί ιδιαίτερη πρόοδος το πρόβλημα της τρομοκρατίας, τα προβλήματα εξωτερικής πολιτικής θα μπορούσαν να λυθούν ευχερέστερα αν ε, ε, σημειωνόταν πρόοδος σε αυτό το τομέα. Τα τελευταία 20-25 χρόνια και μετά τις ε, πρόσφατες εμπειρίες που είχαμε για τη διαχείριση κρίσεων, νομίζω ότι είναι προφανές ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Προσοχή, που δεν προβλέπεται να είναι ευκολότερες οι προκλήσεις που πρέπει να αντεπεξέλθουμε. Ευχαριστούμε η Μαρτίνα Άντερσον. Ευχαριστώ. Την περασμένη εβδομάδα είδαμε μια πολύ σημαντική συμφωνία ανάμεσα στις δύο βασικά κόμματα στην, ε, στο στη Βόρεια Ιρλανδία. Ε, είναι η μοναδική βιώσιμη πολιτική πλατφόρμα για όσους ε, ζουν με τα κοινωνικά επιδόματα ε, και χρειάζονται βοήθεια από το κράτος. Όμως, οι υποχρεώσεις του άρθρου 2 για την, τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το δικαίωμα στην ανθρώπινη ζωή, δεν εξυπηρετούνται από αυτή την συμφωνία. Η Βρετανική κυβέρνηση κάλυψε το στρατό, τους πράκτορες, σε τους πολιτικούς θεσμούς που με συνωμοσία συμμετείχαν και προκάλεσαν δολοφονίες ε, ε, και συνεχίζεται ε, ε, μία συγκάλυψη του, του ρόλου της Βρετανικής κυβέρνησης στη Βόρεια Ιρλανδία. Ο, ο Επίτροπος Μιούσνιακ πρέπει να επιτρέψει στο Μπέλφαστ για να διερευνήσει το ρόλο της Βρετανίας στην σύγκρουση και για να λογοδοτήσει η Βρετανική κυβέρνηση να σταματήσει αυτή η ατιμωρήσία. Επίσης θα πρέπει να συνεργαστεί με τις οικογένειες ώστε να, υπάρχει, να υπάρξει αποκάλυψη έλλειψη των πληροφοριών για αυτές τις δολοφονίες. Σας ευχαριστούμε. Καμπούς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς και εγώ να αποτίσω φόρο τιμή στα θύματα της, του Παρισιού, της Βηρητού, του Μπαμάκο. Η ιστορία διδάσκει ωστόσο ταυτόχρονα, ταυτόχρονα και συγκεκριμένες πραγματικότητες. Πριν από 40 χρόνια, σαν την περασμένη εβδομάδα, πέθανε ο Φράγκο. Τα εγκλήματά του, ωστόσο, ε, ε, μένουν ατιμόρυτα. Πριν από 75 χρόνια δολοφονήθηκε ο αρχηγός του κόμματος μου της Convergentia Καταλούνια, χριστιανός πιστός, ο οποίος έφτασε μόνο και μόνο στην Ισπανία συνελήφθη και του φεκίστηκε το 1938 για την υποστήριξή του για τη δημοκρατία και το καταλανικό έθνος. Η Ισπανική Δημοκρατία και η Ευ... σε συνέχεια πρέπει να ντρέπεται που δεν αποκατέστησε την αξιοπρέπεια στον άνθρωπο αυτό και σε χιλιάδες άλλους καταργώντας τις συνοπτικές δίκες με τις οποίες του φεκίστηκαν περιμένουν οι οικογένειές, τους, οι οικογένειές τους παρακαλώ να καταγραφεί αυτό στα πρακτικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Πίκουλα. Ο Τονίνο Πίκουλα. Ευχαριστώ. Ε, το θέμα της προστασίας των ευρωπαϊκών συνόρων έγινε τις τελευταίες εβδομάδες ένα θέμα προστασίας των πολιτών. Με δραματικό τρόπο τώρα η κρίση ε, αντιμετωπιζόταν ως ανθρωπιστικό ή οργανωτικό ζήτημα. Όμως μετά από τα πρόσφατα γεγονότα στις Βρυξέλλες έχει γίνει ζήτημα ασφάλειας. Η Ευρώπη είναι ε, σε ένα είδος πολέμου, πολιτικού πολέμου. Δεν την έχουν επιτεθεί προωθεί ξένοι στρατοί, αλλά οι ίδιοι πολίτες της κάνουν έναν άγριο πόλεμο εναντίον της. Οι ρίζες αυτού του φαινομένου είναι ε, σε κάποια μορφή κοινωνική παθολογία. Η ο αποκλεισμό από συστήματα, η μη αποδοχή είναι πράγματα που οθούν αυτού του ανθρώπους. Βέβαια δεν γίνονται αυτόματα τρομοκράτες, αλλά η αλληλεπίδραση κοινωνικών και άλλων παραγόντων όπως το μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι αυτά που ασκούν πιέσει όχι σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε όλα τα επίπεδα. Ευχαριστούμε πολύ. Τσάκη. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή τη στιγμή η ξεκάθαρη φιλοδοξία του της διεθνούς τρομοκρατίας είναι το θέατρο των σειράξεων να έρθει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή ειδικά που είναι κοντά στα Χριστούγεννα. Αυτό λοιπόν ε, μας βάζει σε μια δεινή θέση και ανησυχώ που κάποιοι βουλευτές εδώ υποτιμούν το πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση Είμαι σίγουρος ότι οι πολίτες απαιτούν πράξεις από μας. Πρέπει να λάβουμε τις σωστές αποφάσεις αν θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες θα εμπιστεύονται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρέπει να πέσουμε θύματα σε παραδοσιακά πολιτικά ε, παιχνίδια. Το θέμα δεν είναι ποιος θα είναι ο νικητής και ποιος ο χαμένος. Θέλουμε λογικές λύσεις για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση που έχει προκύψει. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει προτείνει ένα πακέτο λύσεων και ο σκοπός αυτών των μέτρων είναι να επαναφέρουμε το αίσθημα της ασφάλειας στους πολίτες. Ζητώ από τους ε, συναδέλφους να ψηφίσουν αυτό το πακέτο γιατί αλλιώς θα φτάσουμε στα πιο ακραία άσχημα φαινόμενα που μπορούμε να φανταστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Κλαούντια Ταπαρτέλη. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης ασφαλείας, η ευρωπαϊκή διαδικασία πρέπει να συνεχίσει. Δεν πρέπει αυτή η κρίση να φτάσει σε εμά. Δεν πρέπει να πέσουμε στην αδράνεια σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης. Πρέπει να συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε τις δουλειές για τους νέους, παρά, παρά το γεγονός ότι συχνά Ξεχνάμε τους νέους και το πόσο ευάλωτοι είναι. Αυτά τα προβλήματα δεν περιμένουν. Επιδεινώνονται. Έχουμε 4,6 εκατομμύρια στην Ευρώπη νέων που δεν έχουν δουλειά. Η Ευρωπαϊκή Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να φέρει ε, περισσότερα στοιχεία σχετικά με τα προγράμματά της ε, που φέρνουν δουλειά στους νέους. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να έχουμε περισσότερες πρωτοβουλίες, μεγαλύτερες επενδύσεις για να μειώσουμε την ανεργία των νέων και γι' αυτό προτείνω αυτά τα προγράμματα να ε, αγγίζουν ανθρώπους μέχρι και 35 ετών. Αυτό το θέμα δεν πρέπει να βγει από την ημερήσια διάταξη και δεν πρέπει να βγει και από τις δημόσιες υπηρεσίες γιατί αυτό το πρόβλημα θα επηρεάζει τις μοίρες όλων μας στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πριν από δύο εβδομάδες εγκρίθηκε η τελική πράξη του Ελσίνκη. Πριν από 20 χρόνια, εδώ στο Στρασβούργο, υπογράψαμε τη Συμφωνία Πλαίσια για την προστασία των ε, μειονοτήτων. Είναι διπλή επέτειο και θα πρέπει να κάνουμε απολογισμό πεπραγμένων και να παραμείνουμε σε γρήγορση, διότι πολλά πρέπει να γίνουν ακόμη για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τα άρθρα που σχετίζονται με την προστασία των μειονοτήτων. Α είμαστε ειλικρινεί. Τα συμβαλλόμενα κράτη δεν εφαρμόζουν πολλά άρθρα της Συμφωνίας Πλαίσιο και θεωρώ θα μπορούσαν να λυθεί αυτό το πρόβλημα εάν ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση μια συμφωνία πλαίσιο για την προστασία των μειονοτήτων. Θα έπρεπε να είναι νομικά δεσμευτική η διάταξη. Την πρωτοβουλία θα πρέπει να την λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμω το Κοινοβούλιο προστατεύει τα συμφέροντα των πολιτών, θα μπορέσει να αναλάβει ηγετικό ρόλο ε, σε αυτό το τομέα. 40 εκατομμύρια ανήκουν σε μειονότητε ε, στην Ευρώπη και το άρθρο 2 τη ε, Διοικητική Λειτουργία Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει ότι η λειτουργία τη Ένωση βασίζεται στην προστασία των μειονοτήτων μεταξύ άλλων. Σα ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Έχουμε μόνο 25 λεπτά χρόνο για να ψηφίσουμε για και να αποφασίσουμε ποιος θα πάρει το βραβείο Λούξ ε, το 2015. Θα απονεμηθεί αύριο το βραβείο στην Ολομέλεια και το αναφέρω αυτό διότι Ορισμένε φορέ ε, η γλώσσα μια κινηματογραφική ταινία είναι πολύ πιο κατανοητή για του πολίτε Ευρωπαϊκή Ένωση από οτιδήποτε άλλο με το Μεντιτεράνια, βλέποντας ε, ε, τα κίνητρα των ε, μεταναστών και προσφύγων από την Αφρική ή επίσης για το ρόλο των μειονοτήτων, τουρκικών μειονοτήτων εδώ στην Ευρώπη. Βλέπουμε λοιπόν ότι ε, ε, ξεκινάει μια συζήτηση για τις ευρωπαϊκές αξίες ε, με αφορμή τέτοιες ταινίε. Πιστεύω ότι το βραβείο Λούξ μας βοηθά να προωθήσουμε τις ευρωπαϊκές αξίες με τον απλούστερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστούμε. τον Ευχαριστώ πρόεδρε. Αυτή την εβδομάδα έπεσε το πρώτο χιόνι σπίτι. Πάμε στο χειμώνα. πολύ. το χειμώνα ξοδεύουν περισσότερα για την ενέργεια. Η ενεργειακή φτώχεια είναι ένα βασικό πρόβλημα. Έχουμε κάνει πρόοδο στη βελτίωση της αποδετικότητας και μείωση του κόστου, ωστόσο τα προγράμματα υποστήριξη από την κυβέρνηση παραμένουν ε, σημαντικά. Η αγορά δεν μπορεί να επενδύσει μόνη τη, ιδίω για όσου μένουν σε εργατικέ κατοικίε. Γι' αυτό η πρόσφατη απόφαση των Τόρις να κόψουν την υποστήριξη για την ε, ε, ηλιακή ενέργεια είναι θλιβερή, γιατί μόνο αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει 26 δις, ε, η επένδυση αυτό μπορεί να είναι 26 δις λίρες και θα ήταν μια σημαντική επένδυση για το μέλλον μας. Ε, δίνοντας χρήματα σε τοπικές κοινωνίες όπως τη δική μου, θα πρέπει να αλλάξει η κυβέρνηση αυτή την, ε, την, την κοντόφθαλμη πολιτική της. Ευχαριστώ. Κλοντ Ρολάου. Παρακαλώ. Το θέμα της αναγνώρισης ε, της, ε, του καθεστώτου της οικονομίας αγοράς ε, στην Κίνα έχει σημαντικές επιπτώσεις για την απασχόληση στην οικονομία μας. Κυρίως διότι η Κίνα ασκεί μια πολιτική επιθετικού χαρακτήρα στα εμπορικά ζητήματα. Αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο στον τομέα της χαλιβουργίας, όπου το, οι ιδιοκτήτες και τα συνδικάτα έχουν τις ίδιες απόψεις. Δεν είναι η οικονομία αγοράς η Κίνα, δεν σέβεται τον, τους κανόνες, τις αρχές του ε, ανταγωνισμού. Οι πρακτικές της θα ήταν επιβλαβείς για εκατοντάδες χιλιάδες θέσεων εργασία άμεσα και ακόμη περισσότερους έμεσα για όλη την οικονομία μας. Η αναγνώρισή της ως μια οικονομία αγορά στην Ευρώπη, η Κίνα πρέπει να πληρεί πέντε τεχνικά κριτήρια. Πόρο απέχει από αυτό. Πρέπει να προσπίσουμε τις αξίες της οικονομίας με κοινωνική ρύθμιση και να μην δώσουμε το καθώς αυτό στην Κίνα. Πρόκειται για θέμα ζωής και θανάτου για το μέλλον της οικονομίας και για το μέλλον της βιομηχανίας μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τελευταίος ο για σήμερα ο κύριος Ιστβαν Ουίχαλη. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι σχεδόν 11 παρατέταρτο. Το βλέπουμε ε, από το ρολόι πάνω από τις ευρωπαϊκές ε, ε, σημαίες και θα είμαι αργός και με υπομονή θα πω αυτό που θέλουν πολλοί να ακούσουν σήμερα εδώ. Όλοι φοβόμαστε τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Οι πολιτικές δυνάμεις χρησιμοποιούνται για την προπαγάνδα κατά των προσφύγων. Όμως, να είμαστε ξεκάθαροι, το πραγματικό πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα εντός της ευρωπαϊκής κοινωνίας και εγώ γι' αυτό θέλω να μιλήσω, για τη φτώχεια των παιδιών. 26 εκατομμύρια παιδιά στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι φτωχά. Ένα στα τέσσερα παιδιά ζει στην ανέχεια στην Ουγγαρία. Είναι τεράστια αυτή η ανισότητα. Μιλάμε ε, για 4,4%. 41,4% ζητώ συγγνώμη. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Αύριο πρέπει να ψηφίσουμε και να δώσουμε ένα τέλος στην παιδική φτώχεια στην Ευρώπη. Οι κυβερνήσει μας πρέπει να λάβουν γνώση αυτού και πρέπει επιτέλους να δώσουν ένα τέλος στην παιδική φτώχεια, να την εξολοθρεύσουν γιατί δεν μπορούμε να έχουμε τίποτα στην Ευρώπη αν παραμένει η φτώχεια στα παιδιά. Ευχαριστούμε κύριε Ουχαή. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να σας πω τώρα ότι αύριο στις 24 Νοεμβρίου θα ξεκινήσουμε στις 8.30 τη συνεδρίαση. Μετά ε, θα υπάρχει ε, μια, μέχρι τις ε, 2.30 και μετά θα ξεκινήσουμε πάλι στις 3 μέχρι τις 11.